Επιτροπή για την παρακολούθηση των αξώνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελευθέρων επαγγελμάτων. Πρώτος ομιλητής, ο συντάκτης της προφορικής ερώτησης, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι βουλευτές, στην Ευρώπη οι τα 4 εκατομμύρια ελευθέρων επαγγελματιών δημιουργούν 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας με κύκλο εργασιών Κύριε Επίτροπε, λίγο ησυχία παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι στην Ευρώπη 4 εκατομμύρια ελευθέρων επαγγελματιών δημιουργούν 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας με κύκλο εργασιών πάνω ε, άνω των 500 δισεκατομμύριων ευρώ. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε για πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε πιστώσει και να μην υπάρχει ε, περιτό γραφειοκρατικό άχθο. Ε, θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίε να χαίρουν των ίδιων ευκαιριών που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Όπω για παράδειγμα πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση από πλευρά ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετοχή στου μειοδοτικού διαγωνισμού και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Μία ομάδα υψηλού επίπεδου που είχα συστήσει όταν ήμουν επίτροπος ε, για θέματα βιομηχανίας το 2014 παρουσίασε μία σειρά από προκειμένου να υποστηρίξουμε το ρόλο των ελευθέρων επαγγελματιών στην Ευρώπη. Όχι μόνο μέσω καλύτερης πρόσβασης πιστώσει, αλλά με περαιτέρω κατάρταση, με περισσότερε πληροφορίε και ε, με ε, γνώμονα την διεθνή του παρουσία. Ήγηκε η ώρα λοιπόν να προχωρήσουμε με αυτές τις ε, ε, προτάσεις και η ομάδα που, έκα, ε, που σύστησα με τη συμμετοχή των διαφόρων πολιτικών ομάδων ρωτά πώς μπορείτε να συνεχίσετε τις δεσμεύσεις που αναλάβετε. Εμείς θα θέλαμε μια ισχυρή δέσμευση από πλευράς της Επιτρόπου Μπιανκόφσκα. Αγαπητή Επίτροπε, σας διαβεβαιώ ότι μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη μιας μεγάλης πλειοψηφίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω νομοθετικών προτάσεων, ε, πρωτοβουλειών και ε, επενδύσεων υπέρ της ανάκαμψης μιας πολύ σημαντικής κατηγορίας στην Ευρώπη. Μια κατηγορία που πρέπει να δει ότι είναι κοντά της ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι' αυτό και απαιτούμε από εσά και περιμένουμε από εσά μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για τα ελεύθερα επαγγέλματα που χρειάζονται περισσότερη ελευθερία και λιγότερη γραφειοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η επόμενη συντάκτρια. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντικά τα ελευθερία επαγγέλματα. Είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επαγγέλματα με υψηλό βαθμό κατάρτισης και δεξιοτήτων. Κυρίως μιλούμε για το, τους ε, τομείς της ε, υγείας, της δικαιοσύνης και άλλους που έχουν να κάνουν με τη δημόσια ασφάλεια και γι' αυτό χρειάζεται υψηλή κατάρτιση. Πρέπει να μεριμνήσουμε για την θέσπιση σαφών κανόνων που θα εξασφαλίζουν την ύψιστη ποιότητα των επαγγελματιών. Συμφωνούμε με τον Σαλφατογιάννη ότι δεν πρέπει να υπάρξει περιττή γραφειοκρατική επιβάρυνση, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε πως έχουμε υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Και ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε. Στον ε, τομέα λοιπόν της ε, εφαρμογής της οδηγίας για τις επαγγελματικές ε, δεξιότητες γίνεται λόγος για μια διαδικασία αξιολόγησης. Ξέρω ότι στους τομείς αυτής, αυτούς γίνεται πολύ προσεκτική εξέταση των δεξιοτήτων. Θα ήθελα λοιπόν μια ερώτηση να μου απαντήσετε. Σε ποιο βαθμό μπορείτε να δώσετε όθηση προς την κατεύθυνση αυτή από τη δική σας από το δικό σας το μετερίζει, πώς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτήν την ε, αξιολόγηση. Γιατί είναι ζητήματα που μας απασχολούν πολύ και όπως είπα, θέλουμε οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους επαγγελματίες αυτούς να προσφέρονται στο ύψιστο δυνατό επίπεδο για τον καταναλωτή, τον ασθενή, για οποιονδήποτε απευθύνεται στους επαγγελματίες αυτούς για να στήσει υπηρεσίες τους θέλουμε τον ύψιστο δυνατό βαθμό εξυπηρέτησης. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκέμπχαρτ και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο έχει η κυρία Μπερνικόφσκα. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να υπογραμμίσω το, τη σημασία και το ρόλο των ελευθερών επαγγελματίων στην Ευρώπη. Πολύ σωστά υπογραμμίζετε ότι έχουν ε, κατά κύριο λόγο επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για δικηγόρους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητες επιχειρήσεις που επενδύουν τα, τους, τα κονδύλια τους και τις γνώσεις τους και χτίζουν την επαγγελματική επιτυχία. Δημιουργούν θέσεις εργασίας και προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναλάβει μια δέσμευση ιδιαίτερα σημαντική για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο σχέδιο δράσης 2020, ενισχύοντας τις, ε, τα ελευθερία επαγγέλματα τον ε, χώρο της ε, τεχνογνωσίας, των δεξιοτήτων, την πρόσβαση στις αγορές που είναι λίγο πολύ ίδια, αλλά ιδιαίτερα δίνουμε έμφαση σε αυτά τα επαγγέλματα. Με μια αυτόνομη ομάδα εργασίας η οποία καταθέτει μια σειρά συστάσεων που περιλαμβάνουμε στην εκθέση την οποία θα δείτε προς το τέλος του έτους και η οποία αναπτύσσεται γύρω από πέντε θεματικές ενότητες. Η πρώτη έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα, γιατί οι επιχειρηματίες αυτοί χρειάζεται να αποκτήσουν και ε, δεξιότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχουν προγράμματα, πρόγραμμα από το οποίο υπάρχει πρόγραμμα από το οποίο μπορούν να αφοληθούν το Εράσμος και τους νεαρούς επιχειρηματίες. Επίσης πρόσβαση σε ε, χρηματοδότηση και σε αυτό θέλουμε ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι προσφέρονται κονδύλια από προγράμματα όπως το COSME, το Horizon 2020, συμβουλευτικές υπηρεσίες του δικτύου Enterprise Europe, τρίτη ενότητα ανάλυση της τα τέταρτη ενότητα πρόσκληση προσώπων από τα ελευθερία επαγγέλματα να ε, συμβάλλουν στο στόχευση της ελάφρυνσης του γραφειοκρατικού φόρτου με, το, τον εντοπισμό είτε των στενοπών είτε των βέλτιστων πρακτικών και πέμπτον ενίσχυση της συμμετοχής των ελευθερίων επαγγελμάτων στην, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, κληθούν, να εκπροσωπηθούν στην Σύνοδο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του 2015 που θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο τον Νοέμβριο εφέτος και εκπρόσωποι των αλευθερίων επαγγελμάτων ώστε να τοποθετηθούν και να ενημερωθούν για όλες τις πολιτικές. Για τα ε, ρυθμιζόμενα επαγγέλματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί σε μία αξιολόγηση διαφάνειας και μηδές αναγνώρισης για όλα τα κράτη-μέλη σε σχέση με την οδηγία των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται σε, στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές πρέπει να πούμε και έχει δώσει στοιχεία σχετικά με 5.000 ρυθμιζόμενα επαγγέλματα σε όλους τους τομείς, σε όλα τα κρατημέλη. Αυτό μας βοηθά ιδιαίτερος γιατί γνωρίζουμε ότι μεγάλη πλειονότητα πλειονότηση των, των ελευθερίων επαγγελμάτων είναι ρυθμιζόμενα. Ε, αυτό συμπέδει και περιορισμό της πρόσβασης και περιορισμό των ευκαιριών για απασχόληση στα ελευθερία επαγγέλματα. Θέλω εν προκειμένου να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σχεδιάζει να υιοθετήσει στρατηγική για την πρόσβαση σε αγορές από τον Οκτώβριο και αυτό σημαίνει περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες και θα διευκολύνει και τις οικονομικές δραστηριότητες των ελευθερών επαγγελματιών. Με χαρά θα συζητήσω περαιτέρω μαζί σας όταν θα είναι έτοιμη και η σχετική στρατηγική το θέμα αυτό γιατί είναι ένα έγγραφο ε, διεξοδικό ευρύ. Έχουμε προσθέσει αρκετά σημεία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ερώτηση αυτή και σας ε, καλώ ε, σε συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστώ την Επίτροπο και τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και πρώτου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Σφάπ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, κυρία Επίτροπε και ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας και την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο βλέπετε το ρόλο των ελευθερίων επαγγελματών στην ιστορική αγορά. Ο Σαν Φωσταζιάννη με πολύ σαφή τρόπο εξήγησε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε εμεί ω Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στου ελεύθερου επαγγελματίε και στα ελευθερία επαγγελματά σε κάθε του εκδοχή. Υπάρχει ανησυχία σε σχέση με ορισμένε διαδικασίε ή παραβάσει κατά κρατών μελών ε, που έχουν να κάνουν με την προστασία των καταναλωτών βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας ότι η κινητικότητα στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά πρέπει να ενισχυθεί οι διαδικασίες αυτές, οι παραβάσει, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στο να διευκρινιστεί αν είναι επιτρεπόμενες αυτές, ε, αυτοί, επιτρεπόμενοι αυτοί οι περιορισμοί από τα κράτη-μέλη ή όχι και γι' αυτό περιμένω να δω και την ετοιμιγωρία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ταυτόχρονα βεβαίως, κυρία Επίτροπε, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει τα ελευθέρια επαγγέλματα, γιατί ως εκ της φύσεώς τους και της αυτοδιαχείρισής τους ε, θα πρέπει, το έχουν αυτό, θα πρέπει να διαφυλάξουν λοιπόν την θέση τους μέσα σε μια ιστορική αγορά και εσείς ως επίτροπος της κλασικής εκδοχής ιστορικής αγοράς εν αντιθέσει προς την ψηφιακή εσωτερική αγορά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσετε τις δικές σας, τις δικές σας εκδοχή της κατάστασης και ιδιαίτερα θα ήθελα να παρελθεύσετε τους κανόνες που αφορούν αυτά τα ελευθερία επαγγέλματα η στρατηγική για την εσωτερική αγορά που θα μας καταθέσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα πιστεύω θα είναι θετική και για τα ελευθερία επαγγέλματα. Ευχαριστώ θερμά. εκ μέρους των Σελιστών και Δημοκρατών. Ο κύριος Δάντη, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει όλο ένα και περισσότερο να βασίζεται στη γνώση ως κινητήριο μοχλό της ανάπτυξή της, ε, τα ελεύθερα επαγγέλματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης παρά το γεγονός ότι την χάνει ελάχιστη προσοχή από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η ανάγκη μεγαλύτερης ε, ένταξης ε, των ελευθερών επαγγελμάτων βάσει συγκεκριμένων και κοινών κανόνων επισημαίνεται και από τα στοιχεία και από την μικρή κινητικότητα των ευρωπαίων επαγγελματιών η μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποδεικνύει αρκετά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να εργαστούμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει το στίχημά μας να είναι η επιμόρφωση και η κατάρτιση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού. Θα πρέπει επίσης να προχωρήσουμε και σε μείωση των ε, ε, γραφειοκρατικών ε, υποχρεώσεων, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και σαφές, ώστε να προσφέρει και ευκαιρίες. Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε και τις δεσμεύσεις της Επιτρόπου που ακούσαμε απόψε για να έχουμε μια ε, κατάλληλη ανάπτυξη αυτής της πολύ σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Ευχαριστούμε κύριε Ντάντη. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, η κυρία Χαράντσοβα για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ε, τα ελεύθερα επαγγέλματα αποτελούν τμήμα της ζωής μας. Θα πρέπει πάντα να την χάνουν σεβασμού και ισότιμων ε, δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώ και η αναθεωρημένη οδηγία είναι τόσο σημαντική. Από του χρόνου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί κάποια επαγγέλματα έχουν εθνικές απαιτήσεις ε, που οποιοδήποτε θα μπορούσε κάλλιστα να σας πει ότι είναι δεν είναι απαραίτητες και αποτελούν διάκριση κατά των ανθρώπων οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρή όταν θα αποφασίζει ποια είναι η δέουσα αιτιολόγηση ε, και να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη που δεν σέβονται το πνεύμα και τις αρχές του νόμου. Κύριε Πρόεδρε, οι Τσέχοι μηχανικοί, οι λογιστές ε, μπορεί να αντιμετωπίζουν μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος όταν θέλουν να ε, μετακομίσουν στη Γερμανία και αυτό σημαίνει ότι ακόμα μας απομένει δουλειά να κάνουμε. Όχι μόνο είναι εις βάρος αυτών των ε, ε, επαγγελματών, αλλά και οι Γερμανοί πολίτες ή και οποιοδήποτε άλλος πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να τους προσφέρονται αυτές οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Ευχαριστώ. Η κυρία Λιγκρίπ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην προηγούμενη θητεία ήμουν συγχύτρια για την εκμέσου ομάδα ΕΛΚ για την αναθεώρηση της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Με αυτό το, μου την ιδιότητα μιλώ σήμερα. Στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, έχουμε καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ε, εφαρμογή της οδηγίας αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Οπότε το διακύβευμα σήμερα σε μεγάλο βαθμό είναι η κινητικότητα των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κινητικότητα αποτελεί ένα από τα κλειδιά για την πρόθεση της ε, ανάπτυξης και της απασχόλησης η αναθεωρημένη η οδηγία περί επαγγελματικών προσόντων ε, επικεντρώθηκε στην ε, χάρτα, την Ευρωπαϊκή Χάρτα Επαγγελματικών Προσόντων που θα διευκόλυνε τις ε, δυνατότητες ε, αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων και επαγγελματιών. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στην κυρία Επιτροπέ, στην ε, υλοποίηση αυτής της επαγγελματικής ευρωπαϊκής χάρτας. Πολλά επαγγελματά ζήτησαν, ενδιαφέρθηκαν να συμπεριληφθούν, οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν για τις νοσοκόμες, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές, ε, τους μεσίτες ε, και μερικά άλλα επαγγέλματα. Πού βρισκόμαστε όμως αυτή τη στιγμή, ε, πόση απόσταση έχουμε διανύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, ο κύριος Σατμάρ Καράς, ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2003 είχαμε Εγκρίνει ένα κοινό ψήφισμα για τους κανόνε ανταγωνισμού και τη ρύθμιση αγοράς ε, για, τα ελευθερία επαγγέλματα. Και μάλιστα για τον απλό λόγο ότι τα ελευθερία επαγγέλματα είναι παράγον τη σταθερότητας σε μια οικονομία. Τώρα βρισκόμαστε ενώπιον νέων προκλήσεων και ιδιαίτερως στην εποχή της ψηφιοποίησης και της παγκοσμιοποίησης. Είναι σαφές ότι τα ελευθέρια επαγγέλματα με ε, πανεπιστημιακά πτυχία και υψηλό επίπεδο ε, δεξιοτήτων κατά κανόνα, ανεξάρτητα, ανεξάρτητοι επαγγελματίες, ουδέτεροι, αντικειμενικοί, αμερόληπτοι, μεριμνούν για την παροχή μιας υπηρεσίας ευραίως φάσματος, δεν μπορούν να ε, να θεωρηθούν δηλαδή ότι είναι κοινοί επαγγελματίες προσφέρουν υπηρεσίες σε τιμές που θα πρέπει να είναι θεμητές σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Όταν μιλούμε λοιπόν για ρύθμιση, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κανόνες οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια, την ελευθερία και την αμεροληψία των ελευθέρων επαγγελματιών. Όχι υπερβολικούς κανόνες, πρέπει να μπορούν να εργάζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίε κατά τρόπο ανεξάρτητο και ελεύθερο. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα ο κύριος Σαλίνη. Ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Επίτροπε. Το θέμα αυτής της ερώτησης άπτεται ενός ε, από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα αλλά ταυτόχρονα και από τα λιγότερα ε, ρυθμισμένα από νομική σκοπιά. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των ελεύθερων επαγγελμάτων ε, εκπροσωπείται ιστορικά πάρα πολύ καλά από τις ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως υπενθυμίζει και η προφορική ερώτηση, ε, έχουμε επισημάνει τις βασικές προτεραιότητες, την ανάγκη της διεθνούς παρησίας, της πρόσβασης στην χρηματοδότηση και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, κύριε Επίτροπε, ε, θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη επαλήθευση του τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μου επί παραδείγματι. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της μορφής με την οποία συνδέονται συχνά ε, τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν αναγνωρίζεται ουσιαστικά. Ε, αναγνωρίζεται τυπικά αλλά όχι ουσιαστικά. Πολύ συχνά αυτές οι ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών έχουν ε, δυσκολίες σε πρόσβαση ε, μορφών χρηματοδότησης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει ανάπτυξη και καινοτομία. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να προσέξετε ιδιαίτερο στο στοιχείο αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σαλίνη. Ο κύριος Σάινφιλτ τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητούμε αυτό το θέμα σήμερα. Τα ελευθερία επαγγέλματα είναι σημαντικά όχι μόνο για την εσωτερική αγορά, έχουν ιδιαίτερη κοινωνική αξία. σε ορισμένε ε, ε, θα πρέπει να περιορίσουμε τους, το κανονιστικό πλαίσιο και σε μερικές περιπτώσεις να το καταργήσουμε για ορισμένα επαγγέλματα. Παρ' όλα αυτά ορισμένα λόμπι ε, και ομάδες πίεσης επηρεάζουν τις κυβερνήσεις και γι' αυτό το λόγο η, η νομοθεσία δεν έχει εφαρμοστεί σωστά ως τώρα πολλές φορές. Πολλές φορές δηλαδή η νομοθεσία περιορίζει την πρόσβαση σε ορισμένα επαγγέλματα εκ μέρους των νέων και αυτό οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας ε, ε, νέων με πάρα πολλά προσόντα. Επίσης επηρεάζει τις τιμές. Οι τιμές παραμένουν υψηλές, ε, δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ελπίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh... Πρόεδρος. Περνάμε στην διαδικασία του Catch the Eye. Τερέσα Κομοντίνη Κάκια. Uh, Δεν ζήτησα το λόγο για αυτό το θέμα, αλλά για το επόμενο, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Okay. Uh... Καλώς. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το λάθος. Ο κ. Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, τα ελεύθερα επαγγέλματα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ένωσης. Όπως ακούσαμε, πάνω από 4 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται στην Ένωση σε σημαντικούς τομείς όπως η υγεία, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια. Ο κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ η οικονομική κρίση όμως έχει χτυπήσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. χρειάζονται λοιπόν μέτρα κυρίως στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσώπων και της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για εξυγχρονισμό του εξοπλισμού τους. στην ελλάδα οι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν χτυπηθεί οικονομικά από το μνημόνιο χτυπιούνται από τη φορομπηκτική πολιτική της τρόικας και χιλιάδες από αυτούς είναι πλέον άνεργοι χωρίς κοινωνική ασφάλιση αλλά και χωρίς να δικαιούνται καν επίδομα ανεργίας. πρέπει λοιπόν να υπάρξουν κοινωνικά μέτρα στήριξης των ελευθέρων επαγγελματιών όχι μόνο στην ελλάδα αλλά και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ένωσης καθώς έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση. ευχαριστώ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ, τον κύριο Μαριά. Και τώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση με την Επίτροπο κυρία Βενικόφσκα. Συγχαρητήρια κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη και τις ε, πολύ λεπτομέρειες ώρες ώρες ερωτήσεις σας Έχω να συμπληρώσω μόνο πως η Επιτροπή αναγνωρίζει το επιχειρηματικό δυναμικό των ε, ελευθερίων επαγγελμάτων και εν προκειμένου θα συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή στα ελευθερία επαγγέλματα στο πλαίσιο, όπως είπα, της επιχειρηματικότητας και το σχέδιο δράσης 2020. Βεβαίως όμως θα συμπεριληφθούν τα ελευθερία επαγγέλματα και στην στρατηγική για την εσωτερική αγορά με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, λιγότερη ε, ρύθμιση. Και επίσης θα κοιτάξουμε με κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις των παραβάσεων, ε, των προσφυγών παραβάση που ανέφερε ο κύριος Ανδρέας Φάπ. Η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από δυνατότητες δράσεις για την αντιμετώπιση των φραγμών που αναφέραν κάποιοι από εσάς όπως δυσανάλογες προϋποθέσεις δεξιοτήτων και κατάρτισης ή υπερβολικές ε, ρυθμίσεις. Το επόμενο θέμα είναι οι αμοιβέ αξιολογήσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων και πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν αφορούν ιδιαίτερα τα ε, ελευθέρια επαγγέλματα. Ο στόχος αυτών των ε, ρυθμίσεων είναι ο περιορισμός των ανάλογα υψηλών φραγμών και των υπερβολικών ρυθμίσεων σε όλα τα επαγγέλματα. Για την αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων, συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα στενά με του εκπροσώπου των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό για να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία για ένα πλαίσιο νομοθετική ε, πράξεω που θα ασχολείται Φερρυπίν για τα, με τα ιατρικά επαγγέλματα. τεχνικές υποδομές και μηχανισμούς ε, του συστήματος πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το 2016 στις αρχές του έτους. Ερώτηση της κυρίας Λεγκρίπ. η δράση που θα ακολουθήσει την αξιολόγηση, αμοιβαία αξιολόγηση θα είναι κομμάτι της ε, στρατηγικής για την εσωτερική αγορά, για την ενιαία αγορά. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί νομίζω θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στο μέλλον να ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά και στην διαδικασία των προσανατολισμών και στην συζήτηση στην Επιτροπή και την υιοθέτηση της ε, στρατηγικής για την εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι έχω πατήσει εν συντομία σε όλες τις ε, ερωτήσεις σας. Κλείνω μόνο λέγοντας ότι ιδιαίτερα θα ενσωματωθούν στη στρατηγική για την ιστορική αγορά τα ελευθερία επαγγέλματα, ο εξυγχρονισμός, ο περιορισμός των ρυθμίσεων, των φραγμών και για τους τομείς αυτούς έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα συνεργαστούμε σας για τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ θερμά.